Λοιπόν, θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ε, το οποίο αφορά στο σχέδιο έκθεση ε, συνοδευόμενο από πρόταση τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο σχετικά με του όρου πιθανή δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού Ιδρύματο για Δημοκρατία. Αυτό ε, είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθότι το θέμα αυτό ε, είναι αντικείμενο πολλών ε, συζητήσεων. Ε, το συζητήσαμε με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Σικόσκι, ε, που εξέφρασε, ο ίδιος εξέφρασε κάποιες αμφιβολίες σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου. Πρέπει να σας πω ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το να έχουμε ένα ευέλικτο αποτελεσματικό ίδρυμα που να προστατεύει τις ε, δημοκρατικές εξελίξεις. Βλέπετε ότι αυτό σήμερα ε, είναι πολύ χρήσιμο. Είδατε ότι προηγουμένως ε, είχαμε δύο πρέσβεις σε ακρόαση τον μελλοντικό επικεφαλής του Σουδάν και τον μελλοντικό επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κονγκό την δημοκρατία του Κονγκό που αποκαλείται δημοκρατία, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι εκεί έχουμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο σε σχέση με ε, την δημοκρατία. Ο συγητής μας είναι ο κύριος Λαμστόφ, ο οποίος θα αναλάβει και την προεδρία όταν θα φύγω εγώ. Έχουμε βέβαια κοντά μας ε, και διάφορους ε, εμπειρογνώμονες και σκιώδεις συντονιστές. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Στανόφσκι, τον Υφυπουργό της Πολωνίας που θα ε, λάβει και εκείνο το λόγο. Θα ήθελα να είσαστε σύντομοι γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Νομίζω όμως ότι θα υπάρξει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και θα ήθελα να ξεκινήσει η κυρία Βαζιλεύσκα η οποία είναι επικεφαλής ε, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για την παρακολούθηση εκλογών και τις δημοκρατικές εξελίξεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πραγματική χαρά για μένα ε, το ότι μπορώ να μιλήσω για αυτό το θέμα. Ε, όπως ε, πολύ καλά γνωρίζετε, έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί στην Νότια Ευρώπη ή μάλλον στις ε, γειτονικές μας χώρες προς νότον. Ε, αλλάζουν συνεχώς λοιπόν οι συνθήκες. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία που να στηρίξει τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού στην περιοχή μας. Και αυτό είναι μία από τις πλέον καινοτόμες ιδέες που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων εξέφρασε την υποστήριξή του για το Ίδρυμα αυτό. Το έπραξε ήδη στα συμπεράσματά του του, ε, της 20ης Ιουνίου και στα συμπεράσματα της προηγούμενης εβδομάδας, της 1 η Δεκεμβρίου, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων εξέφρασε την υποστήριξή του στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία και ζήτησε να υπάρξουν ταχύτατες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Τα κράτη-μέλη συζητούν ε, ένα, μια ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει ε, τα βασικά στοιχεία για ένα Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία. Τα βασικά στοιχεία της ε, έκθεσης συζητήθηκαν ήδη ε, με τις αρμόδιες υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, κυρίως ε, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχει διεξάγει διαβουλεύσεις με, την με κοινωνίες των πολιτών, με ομάδες εμπειρογνωμόνων, γιατί ο βασικότερος στόχος είναι πάνω απ' όλα να υπάρχει ένα εργαλείο σαφούς προστιθέμενης αξίας και συμπληρωματικότητας στα ήδη υπάρχοντα εργαλεία και τις υπάρχουσες πολιτικές. Αναφέρομαι στην πολιτική ε, ανατολική υπάρχουν ε, τα σχετικά ψηφίσματα, αποτελέσματα της απόφασης του Συμβουλίου. Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι λοιπόν οι εξής. Το Ίδρυμα αυτό θα εστιάσει αρχικά την προσοχή του στην, ε, στα θέματα γειτονίας, όμως ε, δεν αποκλείεται στο μέλλον να είναι επίσης ε, σε θέση να ανταποκριθεί σε μεταβατικές διαδικασίες και πολιτικές προκλήσεις σε άλλες περιοχές. Το Ίδρυμα έχει μια σαφή εντολή, είναι ο μηχανισμός χρηματοδότησης πρώτης λύσης για οργανώσεις βάσης συμπεριλαμβανομένων των ε, κινημάτων νέων και για άλλους κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες που δραστηριοποιούνται σε περίοδο μεταρρυθμίσεων. Επίσης ε, θα αποτελεί πηγή στήριξης για όσους αγωνίζονται για τη δημοκρατία. Άρα δηλαδή αυτό που ενδιαφέρει είναι να δημιουργείται δημοκρατικός χώρος ε, με την ελπίδα της μετάβασης. Εδώ λοιπόν το Ίδρυμα αυτό μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο σε σχέση με άλλα ήδη υπάρχοντα ιδρύματα. Το δικό μας αυτό θα είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα. Ε, θα λαμβάνει τις αποφάσεις του ανεξάρτητα, συμπεριλαμβανομένων και όλων των αποφάσεων χρηματοδότησης. Στην ιδανική περίπτωση το ίδρυμα αυτό θα πρέπει να είναι πολύ κοντά ε, στους κοινοτικού ε, θεσμούς. Το ίδρυμα πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις γρήγορα, με ευελιξία. Αυτό λοιπόν είναι το κλειδί, το βασικότερο στοιχείο του Ιδρύματος και αυτό θα έχει ως στόχο να καλύψει το κενό που υφίσταται στα ήδη υπάρχοντα εργαλεία. Γι' αυτό λοιπόν το Ίδρυμα θα έχει ουσιαστική προστιθέμενη αξία. Πάντως, οι κοινοτικοί θεσμοί και κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο θα έχει και μία εποπτεία στη δουλειά του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα θα αναζητήσει τη συνεργασία και με άλλους ε, σημαντικούς εταίρους όπως είναι πολιτικά ιδρύματα, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών για να διασφαλίσει τη συνέπεια, τη συνέχεια αλλά και για να επωφεληθεί από την εμπειρία τους, ε, από την παρουσία τους και για να μην υπάρχουν επικαλύψεις. Το Ίδρυμα θα εκπονήσει κανόνες. Ε, βέβαια, ε, το Ίδρυμα θα πρέπει να διατηρήσει την ισορροπία, αφενός να υπάρχει χρηστή οικονομική διαχείριση, διαφάνεια και λογοδοσία και από την άλλη ε, αποτελεσματικότητα, ευελιξία και ταχεία εκταμίευση πιστώσεων. Όσον αφορά τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σαφές ότι ο κανονισμός, ο σχετικός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνει σεβαστός και θα εφαρμοστεί. Το Ίδρυμα θα χρηματοδοτηθεί καταρχάς ε, σε πρώτη φάση με συνεισφορές των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν στο στόχο, ε, στην αποστολή και στις ε, βασικές αρχές. Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες πρέπει να συμφωνηθούν σε μεταγενέστερη φάση μέσα από τη δουλειά μιας ομάδας εργασίας που θα συσταθεί. Εμείς πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτήν την ομάδα εργασία. Προσβλέπω στι αντιδράσει, ε, τα σχόλια και τι ιδέε σα και είμαι ιδιαίτερα ευτυχή που μπορώ να σα ανακοινώσω ότι ο κύριο ε, Ποπόφσκι θα έρθει και εκείνο κοντά μα ε, γύρω στι 12 και νομίζω και εκείνο θα είναι στη διάθεσή σα για ερωτήσει. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο πρόεδρο, για την πολύ περιεκτική και εμπεριστατωμένη εισήγησή σα και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών τη Πολωνία. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση αλλά και για την θέση που δίνεται στη συζήτηση για τη δημοκρατία και βέβαια για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Δημοκρατία. Στην Πολωνία όταν ε, σκεφτόμαστε για την Ευρώπη, ε, την ε, εννοούμε, την αντιλαμβανόμαστε ως πηγή της δημοκρατίας, ως λίκνο αν θέλετε της δημοκρατίας την περιοχή που ιδρύθηκε η δημοκρατία. Και φυσικά δεν υπάρχει κανένας καλύτερος χώρος για να ε, πούμε και να συζητήσουμε το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τη δημοκρατία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ε, συνένεσης και του διαλόγου στην Ευρώπη. Βέβαια, είναι σαφές ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι σημαντικό να αναζητήσουμε καινοτόμες λύσεις και καινοτόμα εργαλεία. Και όταν ε, μιλάμε για τα οικονομικά ζητήματα, αλλά και όταν ε, εξετάζουμε τις, ξεν, τις διεθνείς σχέσεις, τις σχέσεις μας και με τους γείτονες, αλλά και με τις πιο απομακρυσμένες από εμάς χώρες η ιδέα για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία συζητείται τουλάχιστον το τελευταίο εξάμεινο. Πολλά σχόλια διατυπώθηκαν, εκφράστηκε υποστήριξη, ε, τα κράτη-μέλη διατύπωσαν ε, τις συστάσεις τους και βέβαια και όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συζήτησαν και εξέτασαν τον καλύτερο δυνατό τρόπο λειτουργίας αυτού του Ιδρύματος, γιατί φυσικά μιλάμε για προστιθέμενη αξία η, ε, το κέντρο, ο πυρήνα αυτού του το είναι να αποτελέσει και να προσφέρει προστιθέμενη αξία στις σχέσεις μας με όσους αγωνίζονται για τη δημοκρατία. Με όσους προσπαθούν ε, να έχουν περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες για να αποφασίζουν ε, μόνοι τους για τα θέματα που τους ε, αφορούν. Φυσικά δεν επικεντρωνόμαστε στη Βόρεια Αφρική μόνο και στην Αραβική Άνοιξη. Απλά ε, για μένα αποτελεί μεγάλη τιμή που είμαι εδώ ε, μαζί με τον Βλάντ Βιλίτσκα που είναι φίλος μου στη Λευκορωσία για δύο δεκαετίες, κάτι τέτοιο ε, είχαμε συνεργαστεί προσπαθώντας να οικοδομήσουμε σχέσεις μεταξύ των δημοκρατών της Πολωνίας και των δημοκρατών της Λευκορωσίας. Χρειαζόμαστε αυτό το είδημα για τη δημοκρατία και ε, στην νότια εταιρική σχέση και στην ανατολική εταιρική σχέση, αλλά και σε άλλες χώρες όπως το Μιανμάρ, ε, η Βυρμανία. Ίσως να μην είναι ε, ο μόνος, η μόνη χώρα, αλλά σαν, χώρες σαν αυτές, σαν την, το Μιανμάρ, νομίζω ότι αξίζουν μια ευκαιρία για περισσότερη δημοκρατία. Η Πολωνία σε αυτό το θέμα που αφορά την ίδρυση αυτού του Ταμείου Ιδρύματος για τη Δημοκρατία ε, ακολουθεί ως να τον την, την πιο φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση που μπορεί να ακολουθήσει. Φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίσει έναν ειδικό ρόλο. Όπως βέβαια ε, σημαντικός θα είναι και ο ρόλος της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης για την επιτυχία του εγχειρήματο. Όπως αναφέρθηκε το μέσο αυτό θα πρέπει να είναι γρήγορο, ευέλικτο, αποτελεσματικό και να βοηθήσει στην καθιέρωση του πλουραλισμού και του διαλόγου στις χώρες και τις κοινωνίες αυτές όπου δεν υπάρχει ελευθερία στους τομείς αυτούς και όπου δεν υπάρχει πλουραλισμός. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό να δει κανεί ε, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο Μπουσάν, στην τελευταία σύνοδο της ομάδας υψηλού επίπεδου. Γιατί εκεί είχαμε συζητήσει διάφορα θέματα. Ε, Παραδείγματο χάρη, νέοι δωρητέ, νέοι χρηματοδότε, Ινδία, Κίνα, Βραζιλία τι πρέπει, τι, ποιος πρέπει να είναι ο δικός μας ρόλος. Αυτό συζητήσαμε εκεί. Τι ευθύνη θα έχουμε εμείς και στην οικοδόμηση συνεργασίας με τις γειτονικέ χώρες. Όχι μόνο όμως με αυτές και με τον ευρύτερο κόσμο. Και βέβαια πώς θα εξασφαλίσουμε το σεβασμό στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. και πώς θα στηρίξουμε τα πολιτικά αυτά κινήματα στους διάφορους φορείς οι οποίοι είναι υπέρ της δημοκρατίας και του πλουραλισμού και οι οποίοι φορείς είναι έτοιμοι να συνεργαστούν για την ε, δημιουργία δημοκρατικών επιλογών για τις κοινωνίες των χωρών τους. Έτσι λοιπόν και εμείς συμμετέχουμε και στηρίζουμε την ιδέα της, ε, του Ευρωπαϊκού αυτού Ιδρύματος για τη Δημοκρατία. Θεωρούμε ότι πρέπει να είναι κοινή πρωτοβουλία, δηλαδή και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ και χαιρόμαστε πάρα πολύ που υπογραμμίσατε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζουμε ε, όταν όλο αυτό θα λάβει μια συγκεκριμένη μορφή να φαίνεται κιόλα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει ρόλο προς το συμφέρον όλων. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο ε, στον επόμενο τίκη, τον κύριο Λιαλίτσκα, ο οποίος αναφέρθηκε ήδη και είναι ο πρόεδρος του Διεθνούς Κονσόρσιουμ ε, Μπελαρούς ε, Λευκορωσία, Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε στη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία. Θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου κυρίως δίνοντας το πλαίσιο της Λευκορωσίας και το τι συμβαίνει εκεί στο κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, γιατί συχνά χρησιμοποιείται η Λευκορωσία ως ένα είδος δοκιμής για να δούμε τι θα πρέπει να γίνει για τη στήριξη της δημοκρατίας και των στις κοινωνίες των πολιτών, αλλά πολλά ε, δεν λειτουργούν πάντοτε. <coughs> Όταν μιλάμε για αυτή την ιδέα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Δημοκρατία, εννοούμε ότι από το Δεκέμβριο του 2010 και μετά οι τελευταίες εξελίξεις οδήγησαν στην κατέρευση της ασταθούς απελευθέρωσης και ζούμε τώρα σε ένα ψυχρό εμφύλιο πόλεμο θα έλεγα. Είμαστε σε μια πολύ διχασμένη κοινωνία. Έπειτα έχουμε πολύ σημαντικές τάσεις ε, για περιορισμό των ε, ανθρωπίνων ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ως παράδειγμα να σας δώσω τους νέες νομοθεσίες για την ε, σε δημόσιες συγκεντρώσεις και τη χρήση του διεθνούς χρηματοδότησης που τώρα διέπονται από πολλούς περιορισμούς και για πολλούς από, πολλά από τα συνηθισμένα βήματα στα οποία θα έπρεπε να προβούν οι πολίτες για να ε, φτιάξουν δημοκρατικούς μηχανισμούς μπορεί να ε, υπάρχει ποινική ευθύνη πίσω από αυτά τα διαβήματα. Έπειτα, όλοι οι ανεξάρτητοι φορεί στη Λευκορωσία συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών φορέων καθώ και των ισχυρών ατόμων, δηλαδή συγγραφείς, φιλόσοφοι, μπλόγγερ και άλλοι, ε, θα πρέπει να θεωρηθούν ως η κοινωνία των πολιτών στη Λευκορωσία γιατί είναι κατακαιρματισμένη η κοινωνία οπότε οτιδήποτε είναι ανεξάρτητο θα μπορούσε να ταξινομηθεί ως κοινωνία των πολιτών. Έπειτα, θα πρέπει σαφώς να κατανοήσουμε πως η κοινωνία των πολιτών έχει περιορισμένη πρόσβαση στον λαό, στον απλό πολίτη. Είναι η αδυναμία, αλλά είναι και η πραγματικότητα που έχουμε. Ε, μια άλλη αδυναμία είναι η έλλειψη επικοινωνίας και συντονισμού ανάμεσα σε δύο μεγάλα τμήματα των ανεξάρτητων δυνάμεων, πολιτικών και κοινωνίας των πολιτών. Ε, έλλειψη, παρεξήγηση, ε, προσπαθούν να οικοδομήσουν την εμπιστοσύνη, αλλά πόρο απέχουμε από αυτό που χρειαζόμαστε. Και κάτι ακόμα όσον αφορά τους πόρους. Μόνο η διεθνή χρηματοδότηση είναι διαθέσιμη όσον αφορά την χρηματοδότηση των δημοκρατικών δυνάμεων στη Λευκορωσία. Εσωτερικοί πόροι δεν υπάρχουν για να χρησιμοποιηθούν για τέτοιου είδους δουλειά. Και η κοινοτική χρηματοδότηση ε, αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, ωστόσο ένα μικρό τμήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εκδημοκρατισμό, γιατί τα προγράμματα όπως ΜΚΟ και τοπική αυτοδίκηση χρειάζεται μικρή χρηματοδότηση για τους φορείς κτλ. Ε, αυτό που ήταν καλό τα τελευταία χρόνια ήταν η πρωτοβουλία Ανατολική Εταιρική Σχέση που έδωσε μια νέα δυναμική στην ε, κοινωνία των πολιτών. Έφερε επίση την πίστη πω είναι δυνατόν να αλλάξουν τα πράγματα και δόθηκε και ευκαιρία για οικοδόμηση σχέσεων με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τουλάχιστον επί τη βάση του φο... της υποδομής του Φόρουμ για την Κοινωνία των Πολιτών. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, τι μας, ε, βρίσκει... τι μας αρέσει στην ιδέα αυτή για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία. Καταρχήν, η ιδέα να συγκεντρωθεί η εντολή αυτού του Ιδρύματος στα θέματα εκδημοκρατισμού, γιατί οι τοπικές αρχές μπορεί να κάνουν παρόμοια πράγματα, αλλά είναι προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Ε, η διευκόλυνση, το μέσο για την ε, δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρόσφατα δημιουργήθηκε ε, Ωστόσο, χρειάζεται μια ευρύτερη δράση σε ευρύτερη κλίμακα. Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία έχει τις δυνατότητες να στηρίξει καινοτομίε. Αλλά και όχι μόνο τυποποιημένες λύσεις. Σε μια χώρα σαν τη δικιά μου χρειάζονται καινοτόμες λύσεις, γιατί οι στάνταρ λύσεις δεν λειτουργούν, τουλάχιστον σε αυτή την προδημοκρατική φάση. Και το Ίδρυμα μπορεί να συμβάλλει σε αυτό. Τρίτον, ταχεία και ανεξάρτητη δράση που χωρίς γραφειοκρατική διαδικασία και λήψη αποφάσεων καθώς και καλύτερη στοχοθέτηση, αυτό που αναμένουμε από το Ίδρυμα, αυτή είναι η, θα ήταν ε, προστιθέμενη αξία, ε, δηλαδή επιπλέον και όχι σε αντίθεση με άλλους μηχανισμούς. Κάτι ακόμα που θα θέλαμε είναι η ιδέα πίσω από το Ίδρυμα, τουλάχιστον για την ώρα αυτό περιγράφεται, είναι ότι δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στους εσωτερικούς φορείς ε, γιατί μόνο ενισχύοντας τις τοπικές ε, δυνάμεις μπορεί να έχουμε αλλαγές. Δεν λέω τώρα ποιες συγκεκριμένες ε, δυνάμεις πρέπει να ενισχυθούν, αλλά αυτέ μπορούν να αγωνιστούν για δημοκρατικές αλλαγές. Ποιε είναι λοιπόν οι προκλήσεις, Ποιε προκλήσεις μπορούμε να εντοπίσουμε για το Ίδρυμα. Περισσότερη χρηματοδότηση για εκδημοκρατισμό σε χώρες όπως η δική μου δεν σημαίνει απαραίτητα και περισσότερη δημοκρατία, δεν είναι άμεση η σχέση. Το θέμα είναι πώς θα επιτευχθεί πρόοδος και ίσως και να είναι αυτό το πιο δύσκολο. Δεύτερον, αν μιλάμε για στήριξη των δημοκρατικών δυνάμεων, ποιες είναι αυτές πώς ε, να εντοπιστούν αυτές σωστά, ποιο είδος υποστήριξη χρειάζονται πραγματικά και πώς να οργανωθεί αυτή η στήριξη με τρόπο ώστε να ενισχυθούν οι δημοκρατικοί φορείς της χώρας. Κάτι ακόμα, μια ακόμα μεγάλη αλλαγή που νομίζω σαφώς την είδαμε πέρυσι για περιπτώσεις όπως ο άλλος Λιάσκη τι να κάνουμε στο θέμα και στο δίλημα μάλλον ανάμεσα στην ε, διαφάνεια και την ασφάλεια. Γιατί εμεί θέλουμε να ασφαλίσουμε τους φορείς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ε, στήριξη από το Ίδρυμα στο μέλλον. Δυστυχώ όμως υπήρξαν περιπτώσεις όπου δεν είμαστε βέβαιοι για την ασφάλεια διότι υπάρχει πολύ διαφάνεια. Συγκεκριμένη δημοκρατική κανόνας που είναι φυσιολογική για την Ευρώπη και για τις δημοκρατικές αρχέ στη Λευκορωσία θα θέλαμε να υπάρχει αυτή η διαφάνεια αλλά η παρενέργεια είναι ότι οι δημοκρατικοί φορείς έρχονται σε δύσκολη θέση και ε, κινδυνεύουν. Πρέπει να βρεθεί λύση λοιπόν γι' αυτό. Αν υπάρχουν προτάσεις που να μπορούν να είναι βοηθητικές από τη δική μας προοπτική, ε, μπορώ να σας αναφέρω ε, τις εξής. Πρώτον, εισαγωγή αρχών διευθυντικού διαλόγου η δημιουργία ενός συστήματος συντονισμού με τους τοπικούς φορείς αλλαγής σε όλα τα επίπεδα από τις αρχικές έρευνες μέχρι τη δημιουργία προγραμμάτων, την εφαρμογή τους και την αξιολόγησή τους. Πιστεύω πως ε, το Ίδρυμα θα είναι πολύ πιο σωστό και στοχοθετημένο αν αυτή η αξιολόγηση γίνεται τακτικά και οι τοπικοί φορείς δεν ε, θεωρούνται μόνο ως δικαιούχοι Δεύτερον, είναι απαραίτητο να οριστούν κριτήρια για την επιλογή των ε, φορέων που θα υποστηριχθούν και καταστάσεις όπου η βοήθεια αυτή είναι απαραίτητη. Η στήριξη, η βοήθεια δεν θα πρέπει να προωθεί την αποσύνθεση των δημοκρατικών παικτών, ούτε να προκαλεί ανταγωνισμό μεταξύ τους, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ αρνητικό και πιστεύουμε, είδαμε μάλλον τέτοιες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της ανατολικής ε, εταιρική σχέσης, όχι ως τμήμα της πρωτοβουλίας, αλλά ήταν μέσα στη δυναμική. Στη Λευκορωσία ε, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη ανάμεσα στην πολιτική, στους πολιτικούς κύκλους και την κοινωνία των πολιτών, ενώ στην Αρμενία υπήρχε πραγματικός ανταγωνισμός ανάμεσα στις διάφορες οργανώσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών. Να αναφέρω και την ιδέα που αναφέρθηκε στην ε, ενημέρωση πολιτικής Φρίντε Μου άρεσε η ιδέα των τριών πυλώνων που στοχεύουν στην ε, προμεταβατική περίοδο, τη μεταβατική περίοδο και την μεταμεταβατική περίοδο. Έτσι θα είναι πιο συγκεκριμένοι οι στόχοι τα και τα προγράμματα και έτσι τελικά θα έχουμε περισσότερα ωφέλη. Τελευταία μου παρατήρηση είναι η ιδέα της συμπερίληψης των ε, βασικών δημοκρατικών εκπροσώπων των υποστηριζόμενων χωρών μέσα στην ε, δομή του Ιδρύματος. Θα μπορούσε να είναι κάποιο είδος συμμετοχή ε, σε διαβουλεύσεις, κάποιο είδους συμβουλευτικό σώμα αν δημιουργηθεί κάποιο συμβούλιο εμπειρογνωμόνων ή κάποια ομάδα εμπειρογνωμόνων πάντως να είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί στην ε, σύνθεση την ίδια του Ιδρύματος. Ευχαριστώ πολύ για τα δύσκολα θέματα που θέσατε αλλά και για τις προτάσεις σας και φυσικά σας ευχαριστώ γενικότερα εξ ονόματος του Κοινοβουλίου για τη σημαντική σας δουλειά. Και τώρα θα ρωτήσω την ε, κυρία Χέιλ πριν δώσω το λόγο στον ε, κύριο Λάμστορφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας κάλεσε να μιλήσουμε εδώ στην Επιτροπή σας. Έχουν υποθεί αρκετά, άρα θα κάνω ό,τι μπορώ για να είμαι σύντομη. Εκπροσωπώ ένα ίδρυμα με τρικονταετή εμπειρία σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών σε πάνω από 70 χρόνια ε, χώρες. Στηρίζουμε τις ε, τοπικές οργανώσεις, ε, τη συμμετοχή τους στις διάφορες διαδικασίες. Πώς, ποια είναι η αφετηρία μας ό,τι αφορά αυτό το είδαμε για τη δημοκρατία. Πριν από κάποιους μήνες αρχίσαμε να ασχολούμαστε αυτό το θέμα και κυρίως μας απασχόλησε η προστιθέμενη αξία. Ακούσαμε και άλλοι να αναφέρονται στην προστιθέμενη αξία. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά μέσα, πολλά ιδρύματα, τα οποία κάνουν πολύ καλή δουλειά στον τομέα της δημοκρατίας και των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Πρέπει λοιπόν το Ίδρυμα για τη Δημοκρατία να έχει κάποια απτήσιμη συνεισφορά στις προσπάθειες αυτές. Ακούσαμε τις προτάσεις της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Εμείς στηρίζουμε ε, το Ευρωπαϊκό Δρόμο για τη Δημοκρατία γιατί θεωρούμε ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας της ευρωπαϊκής υποστήριξης που θα είναι πιο καλά προσαρμοσμένη στους τοπικούς φορείς ε, που θέλουν να προωθήσουν τη δημοκρατία στις κοινωνίες τους. Σήμερα θα αναφέρω πέντε βασικές αρχές που νομίζω ότι μπορεί να ακολουθήσει και το Ίδρυμα για τη Δημοκρατία. Πρώτα απ' όλα, ανάγκη να μπορεί κανείς να αποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες, στα τοπικά ε, θεματολόγια. Είναι μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Δεν τη βλέπουμε συχνά ε, στη στήριξη που παρέχει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν δει κανεί τώρα τι γίνεται στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή, ε, τίθενται ιδιαίτερα θεμητά ερωτήματα. Υπάρχουν τοπικές ευαισθησίες για το ρόλο των εξωτερικών φορέων. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά ε, τις κυβερνητικές δυνάμεις, αλλά και τους ακτιβιστές, τους πολίτες ε, που κάποιες φορές νομίζουν ότι η Ένωση στηρίζει τα παλιά καθεστώτα. Δεν θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να γίνονται στο τίμημα της τοπικής νομιμοποίησης αυτής της στήριξης. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν να βρει μια ισορροπία το Ίδρυμα και να είναι ε, να ακολουθεί τις στρατηγικές ε, αυτές προσεγγίσεις και προτεραιότητες, αλλά θα πρέπει να ακούει και τις ιδέες που προέρχονται από την τοπική κοινωνία. Παραδείγματο χάρη, μέσω διαγωνισμών ανοιχτών και ε, προσκλήσεων υποβολή προτάσεων θα καταφέρει πολύ περισσότερα το Ευρωπαϊκό Αυτοδήμα παρά να βασίζεται στου γραφειοκρότε των Βρυξελών για να κάνουν τι ε, προτάσει και μετά να χρηματοδοτεί τις διάφορες αποφάσεις όπως ισχύει μέχρι τώρα. Δεύτερον, θα πρέπει να στηρίξει διάφορους τομείς που προωθούν τις κοινωνικές αλλαγές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το παρελθόν ε, πολλές φωνές, ισχυρές φωνές ήρθαν από το εξωτερικό και όχι μέσα από τα, ε, τα βασικά παγιωμένα πολιτικά κόμματα. Και πρέπει να το έχουμε υπόψη μα ε, όταν θέλουμε να χαράξουμε αυτό το νέο ίδρυμα. Θα πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν νέου ηγέτε, ε, τα κοινωνικά κινήματα, τα συνδικάτα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επειδή μιλάμε για προσθέμενη αξία, αυτέ οι ομάδε αυτή τη στιγμή δεν ωφελούνται άμεσα από τα εφιστάμενα μέσα. Παραδείγματο χάρη, υποστήριξη στο πλαίσιο του Ιδρύματο θα μπορούσε να έχει τη μορφή υποτροφιών ε, που θα μπορούσαν κάποιοι αντιφρονούντε να έρθουν στην Ευρώπη, να μελετήσουν τι δημοκρατικέ διαδικασίε. Επίσης θα μπορούσε να παρασχεθεί στήριξη στη διασπορά, στα μέσα επικοινωνίας, ε, σε, διάφορους, ε, ε, σε διάφορες ομάδες προβληματισμού, think tanks. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια πρέπει να είναι αμερόληπτη, γιατί στόχος είναι να παράσχει στήριξη στα δημοκρατικά συστήματα και όχι να υποστηρίζει τους νικητές. Δηλαδή δεν θα πρέπει να ε, πρόσκειται ιδεολογικά κάπου. Πρέπει να είναι μη διακριτική η στήριξη που θα παρέχει. Αν παραδείγματο χάρη είχε στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα συγκεκριμένο κόμμα στην Αίγυπτο του τελευταίου μήνε, απλά και μόνο για ε, να γίνουν γρήγοροι όλε οι διαδικασίε και αυτό το κόμμα τελικά δεν το δεχόταν ο λαό τη Αιγύπτου, θα ήταν καταστροφή. Πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικέ δικλείδε και στην οργανωτική δομή. Ε, εκ περιτροπή ε, ε, συμβούλιο από του κυβερνήτε, για παράδειγμα. Εμεί το έχουμε χρησιμοποιήσει αυτό ως δομή για να αποφύγουμε τι συγκρούσει συμφερόντων και για να προωθήσουμε την διαφανή λήψη αποφάσεων για τα σχέδια που πρέπει να τύχουν υποστήριξη. Τέταρτον, είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή στο μεταβατικό πλαίσιο και εδώ μιλάμε κυρίω για μια γραμματεία του Ευρωπαϊκού Δρόμου για τη Δημοκρατία που θα συνεργάζεται με την Εκτελεστική Επιτροπή και θα ξέρει την περιοχή και θα μπορεί να θέτει τα σωστά ερωτήματα για να στηριχθούν οι σωστέ παρεμβάσει. Ακούσαμε από τον προλαλήσαντα τους τρεις πυλώνε να μας αναφέρει των διαφόρων μεταβατικών αυτών περίοδων. Δεν ξέρω αν ε, είναι συγκρίσιμη κατάσταση με τη Γεωργία ή τη Ρωσία. Ε, είναι μετασυγκρο... Ε, κατάσταση ή περίοδος μετά από μία σύγκρουση όπως τη Λιβύη. Τι ακριβώς ισχύει σε κάθε περίπτωση. Τέλος, Ακούσαμε από προηγούμενους ομιλητές ε, να αναφέρονται λέξεις ευελιξία, ανάληψη κινδύνου, καινοτόμος. Αυτά είναι επίθετα που δεν χρησιμοποιούνται σωστά από εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών οποτεδήποτε μιλούν για υπάρχοντα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν μιλήσετε μαζί σας θα καταλάβετε πολύ καλά τι εννοώ. Εμάς ε, μας αρέσει η ιδέα του να υπάρχει ένα εργαλείο πρώτης καταφυγής αντί τελευταίας. Και εδώ συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι είναι μια πρωτοβουλία που μπορεί να ενεργοποιήσει και άλλες ε, ή αν θέλετε και συνεργασίες και άλλα, να κινητοποιήσει άλλα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το Ίδρυμα μπορεί να συμπληρώνει το έργο του Ινστιτούτου Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό. Ε, βεβαίως, ε, ε, πρέπει να είναι κοντά, να βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο και οι ακτιβιστές πρέπει να αισθάνονται ότι αυτό το Ίδρυμα συνδέεται αλλά δεν ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και για τα κράτη-μέλη ε, είναι σημαντικό οποτεδήποτε γίνεται αναφορά από τα κράτη-μέλη σε υποστήριξη της δημοκρατίας να μπορούν οι κυβερνήσεις ε, να καταφύγουν σε αυτό το Ινστιτούτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και προσβλέπω στη συζήτηση. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε και εμείς και ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει αυτό το Ινστιτούτο Θαύμα αν εκπληρωθούν όλα τα κριτήρια, αλλά εν πάση περιπτώσει ας ξεκινήσουμε φλόδεξα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να παραδώσω και το λόγο και την Προεδρία στον κύριο Λάμπστοφ που είναι εισηγητής αυτής της Επιτροπής. Εγώ ε, είμαι σκιώδης εισηγητής ε, και ελπίζω άλλοι να εκφράσουν επίσης ε, τα σχόλιά τους. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε μία επικοδομητική συζήτηση. Η ε, Πολωνική και η Δανική Προεδρία ελπίσουμε ότι θα υιοθετήσουν όλες μας τις προτάσεις και θα έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε το Ίδρυμα γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο όχι μόνο για τις χώρες αλλά για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Λάμπστοκ. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω καταρχήν ευχαριστώντας τους προσκεκλημένους μας που ήρθανε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να ακούμε την άποψη των ανθρώπων που κάνουν επιτόπου τη δουλειά. Και νομίζω ότι είναι επίσης σημαντικό ε, να εντοπίσουμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε στο μέλλον. Ε, ευχαριστούμε λοιπόν τους ε, παριστάμενους, όλους τους παριστάμενους. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις εισηγητές για τις προτάσεις τους μέχρι τώρα, για την επικοδομητική τους προσέγγιση. Και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους από τις Επιτροπές Ανάπτυξης και Γυναικείων Υποθέσεων, γιατί και αυτοί τοποθετήθηκαν και κατέθεσαν προτάσεις τις οποίες ε, θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε υπόψη μας ε, στη διάρκεια όλων αυτών των διαδικασιών που θα ακολουθήσουν. Τις απόψεις μου ε, θα θα τις χωρίσω σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος, γιατί συζητάμε για την ύπαρξη ενός τέτοιου ιδρύματος. Δεύτερον, θα καταθέσω τις βασικές μου προτάσεις και τρίτον ε, θα μιλήσουμε για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μελλοντικές εξελίξεις και σε σχέση με τη λειτουργία του Ιδρύματος. Ξεκινάω λοιπόν υπενθυμίζοντά σας γιατί μιλάμε για αυτό το πράγμα. Είπαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, είναι καλά, δεν ήταν καλά προετοιμασμένη να στηρίξει ε, τους παράγοντες κυρίως ε, κατά την Αραβική Άνοιξη ε, και αναφέρθηκε ότι προέκυψε και κάποια απογοήτευση όσον αφορά στην ικανότητα των δικών μας των θεσμών να ανταποκρίνονται στις ε, αλλαγές που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή στη νότια γειτονία μας. Υπάρχει λοιπόν εδώ κάποιο περιθώριο βελτίωσης ε, κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε την αξιοπιστία μας ε, όσον αφορά αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται, αγωνίζονται για τη δημοκρατία. Βέβαια πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τους περιορισμούς που υπάρχουν ε, σήμερα. Εμείς θέλουμε το Ίδρυμα να είναι μια οντότητα που θα αντιδρά με μεγαλύτερη ταχύτητα, με λιγότερη γραφειοκρατία. Και θέλω να το καταστήσω απόλυτα σαφές ότι δεν μας ενδιαφέρει να ε, αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε εργαλείο ούτε να υπάρχει επικάλυψη εργασιών, κυρίως όχι με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το EIDHR, το οποίο κατά την άποψή μας έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ε, και συνεχίζουμε να το στηρίζουμε. Βέβαια, αυτό έχει περιορισμένη εντολή και αρκετά ε, χρονοβόρες ε, διαδικασίες. Πρέπει λοιπόν και αυτό να γίνει ε, πιο ευέλικτο. Παρ' όλα αυτά όμως το EIDHR θα είναι κάτι διαφορετικό από το δικό μας το Ινστιτούτο και έτσι είναι το σωστό. Πιστεύω ότι το Ίδρυμα αυτό θα προσθέσει αξία στον εκδημοκρατισμό και νομίζω αυτό αναφέρθηκε και προηγουμένως ότι υπάρχει και το σχετικό αίτημα. Ας δούμε λιγάκι ποια είναι τα βασικά στοιχεία της σύστασης. Όπως είπα και προηγουμένως, ε, να υπάρχει συμπληρωματικότητα με τα υπάρχοντα προγράμματα. Επίσης, ένα τέτοιο ίδρυμα θα πρέπει να προσφέρει ευέλικτες, ε, έγκαιρες απαντήσεις και βοήθεια, να προσφέρει βοήθεια στη βάση και να υπάρχει και η δυνατότητα ε, να τροποποιεί τα προγράμματά του θα πρέπει να λειτουργεί σε περιφερειακό επίπεδο, <clears throat> να συγκεντρώνει τεχνογνωσία και να συντονίζεται με τα Ινστιτούτα εδώ ε, στις Βρυξέλλες, κυρίως με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Για μας λοιπόν είναι σημαντικό το Ίδρυμα αυτό να εγκατασταθεί στις Βρυξέλλες. Πρέπει λοιπόν να προσφέρει άμεσες πιστώσεις στους ε, δικαιούχους αποδέκτες, ε, Στόχος είναι μια ευρία ομάδα επίδοξων αποδεκτών συμπεριλαμβανομένων και άλλων σημαντικών παραγόντων όπως ε, κινήματα, ε, νεόκοπα κόμματα, ε, bloggers, ομάδες ανεφρονούντων και το καθεξής. Άρα δηλαδή οι αποδέκτες θα είναι πάρα πολλοί. Επίσης θέλω να σας πω ότι ε, δεν θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει και συγχρηματοδότηση. Η δομή του είναι πολύ σημαντική. Νομίζω το Ίδρυμα αυτό ε, θα έχει έτσι μια υβριδιακή δομή με την έννοια ότι θα είναι μια οντότητα που επιδιώκει την ισορροπία ανάμεσα στην αυτονομία του και τη λογοδοσία. Αυτό είναι καθοριστική σημασία. Και Αν ληφθούν υπόψη αυτά που ανέφερα προηγουμένως, νομίζω ότι το εργαλείο αυτό θα είναι πιο αποτελεσματικό. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να περτώ σύντομα στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ είμαι πεπισμένος για την ε, ισορροπία που μόλις σας περιέγραψα και που μπορεί να επιτευχθεί με τη δική μας τη βοήθεια. Η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ισχύει βεβαίως σεβόμενη όλοι του κανόνες. Εμείς θα πρέπει να έχουμε μια γενική εικόνα, μια εποπτεία όσον αφορά τι δραστηριότητε του Ινστιτούτου. Και το είπα αυτό όχι για θεσμικούς λόγους, αλλά λόγω του ότι εδώ ε, έχουμε πολλούς ε, δημοκρατικά εκλεγμένους βουλευτές που ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει δημοκρατία. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι να συμπεριληφθούν στο μελλοντικό ε, διοικητικό συμβούλιο Ευρωβουλευτέ, αυτό θα βοηθήσει στο να οριστούν οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές του Ινστιτούτου. Βεβαίως ε, πρέπει να δούμε λιγάκι πώς ε, ε, το Ίδρυμα αυτό θα αναφέρεται στην Εκτελεστική Επιτροπή. Τέλος, ε, πιστεύω ότι όλα αυτά ε, θα προσφέρουν στη διαφάνεια και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράκης ανακοίνωσε ότι και το Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει στην ομάδα εργασίας ε, στην οποία θα συμμετέχουν οι Κομισιόν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ελπίζω λοιπόν ότι η σημερινή ακρόαση θα καταστήσει σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να συμμετάσχει επικοδομητικά ε, στο, στο θέμα του Ινστιτούτου και γι' αυτόν το λόγο εξάλλου συστήσαμε και αυτό το σχέδιο συστάσεως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα ε, θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές των διαφόρων πολιτικών ομάδων, εκ των οποίων κάθε ένας έχουν, έχει δύο λεπτά ε, στη διάθεσή του. Ο πρώτος ε, αντικαθιστά ένα συνάδελφο από το ΕΛΚ που δεν μπορούσε να είναι εδώ ε, και δίνω το λόγο στον κύριο Πέτερινγκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Λάμπστοφ, τότε αντικαθιστώ την κυρία Ζαΐφη, το πληροφορήθηκα μόλις από εσάς. Δεν ξέρω όμως αν θα πω ακριβώς αυτά που θα ήθελε να πει η κυρία Ζαΐφη. Έχω την εντύπωση ότι ε, έχει προχωρήσει η διαδικασία. Εγώ δεν θέλω να τοποθετηθώ κατά αυτού του εγχειρήματο, αλλά έχω κάποιες ερωτήσεις. Βεβαίως ε, και είμαστε όλοι μας υπέρ της ε, προαγωγής της δημοκρατίας και έχοντας εδώ φίλους από τη Λευκορωσία ή τέθηκε το θέμα της Αραβικής Άνοιξης. Εγώ έχω πάει σε όλες αυτές τις χώρες και στη Λευκορωσία. Βεβαίως και όλοι μας είμαστε υπέρ της ενίσχυσης της δημοκρατίας. Όμως πρέπει να διερωτηθούμε, έχουμε στα χέρια μας τα απαραίτητα εργαλεία. Ε, κύριε Πρόεδρε, εσείς ε, αναφερθήκατε και είπατε σε αυτό το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημοκρατίας και ότι αυτό ε, έχει δοκιμαστεί στην πράξη και είναι επιτυχές. Τότε γιατί δεν το αναθέτουμε σε αυτό, δεν αναθέτουμε σε αυτό το Ίδρυμα τα θέματα της δημοκρατίας, αλλά επιλέγουμε μία, ένα νέο Ινστιτούτο. Το κάνουμε γιατί ε, πιστεύω ότι θα είναι διακυβερνητικό ε, το Ινστιτούτο. Εκείνο όμω που τίθεται επιτάπτωση είναι ποιο θα ασκεί τον έλεγχο. Με μεγάλη μου χαρά άκουσα ότι ο Κόμι Λάμστοφ πρότεινε τον έλεγχο να τον ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμω ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχο νομίζω από αυτού ε, δεν, έχει, δεν αμφιβάλλει κανεί. Και κατόπιν το ερώτημα ποιο θα είναι αποδέκτης των κονδυλίων, της ενίσχυσης. Είναι σαφές, αποδέκτες θα είναι η κοινωνία των πολιτών ε, στα διάφορα κράτη, αλλά προτείνω και αν μου το προτείνετε αυτό ως ε, πρόεδρος ενός Ιδρύματος Γερμανίας, του Ιδρύματος Κόνετ Αντενό, να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά Ιδρύματα στη Γερμανία. Και ακούσαμε μια έκθεση ε, για εμπειρία που έχει συγκεντρωθεί από διάφορες χώρες η εμπειρία αυτή μας οδηγεί στο να πιστεύουμε ότι το Ίδρυμα αυτό δεν πρέπει σίγουρα να αποκλειστεί. Ε, η δικιά μας η δουλειά του Κοινοβουλίου είναι αυτό το εγχείρημα να λάβει συγκεκριμένα σάρκα και οστά. Και όσον αφορά στις ε, αρχές ε, αυτού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Δημοκρατίας, οι προϋποθέσεις ε, που πρέπει να πληρούνται, αυτές πρέπει να ε, επηρεαστούν, να οριστούν από εμάς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Πέτερινγκ. Ε, θα πράξουμε αυτό που μας συστήνεται και επόμενη είναι η κυρία Βερονίκ Ντεχάιζα που ομιλεί εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών και δεν αναπληρώνει κανένα. Μιλάει εξ ονόματός της. Μάλιστα, κανένα δεν αντικαθιστώ, ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Ισηγητά. Ε, την στήριξη που εν γέννη δίνουν οι ομάδες σε αυτή την ιδέα. Δηλαδή δεν τολμώ να μιλήσω για μέσο, αλλά αυτή την ιδέα να υπάρχει κάτι το οποίο να είναι πιο ευέλικτο που θα μπορεί να χρηματοδοτήσει αναδυόμενους φορείς σε χώρες όπου είναι σε δημοκρατική μετάβαση, σε μεταβατική περίοδο, κατά τη διάρκεια αυτής και μετά. Βλέπω όμως κάποιες ελλείψεις. Υπάρχουν πολλά μέσα και πολλά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας ήδη, ε, ε, ε, αλλά βεβαίως συμμερίζομαι και τις διάφορες προειδοποιήσεις των συναδέλφων και κυρίως του κυρίου Πέτερινγκ για τις πιθανές επικαλύψεις και για τον ακριβή ορισμό του τι θέλουμε. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω στα εξή ε, σημεία και ορισμένα ήδη τα έχουμε κάπως αναφέρει. Πρώτο, εφόσον πρόκειται εν μέρη για ευρωπαϊκά χρήματα και για αρμοδιότητες τις οποίες ασκούμε, ποιος θα είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου θα το βάλουμε στην δομή μέσα, θα μπορέσουμε να κατευθύνουμε τους ε, προσανατολισμούς και να ελέγξουμε μετά τη χρήση των πόρων. Αυτό είναι το μήνυμα. Αλλά στο ρόλο του Κοινοβουλίου θα ήθελα να υπάρχει και μια ε, πολιτική ισορροπία. Δηλαδή το Κοινοβούλιο αποτελείται από πολιτικές ομάδες ε, και θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να υπάρξει μια στάθμιση των πολιτικών ομάδων. Κάτι το οποίο να μην είναι βαρύ, αλλά είναι βασικές δημοκρατικές προϋποθέσεις. Για το θέμα των επικαλύψεων, να, θα ήθελα τα μέσα που υπάρχουν να μην αποδυναμωθούν ούτε μέσω της επικάλυψης, ούτε ε, μέσω των χρημάτων που θα μπορούσαμε να τους ε, πάρουμε. Αν υπάρχουν χρήματα από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, θα ήθελα να ξέρω από πού θα προέλθουν. Αν πρόκειται να τα πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα ενισχυθεί αυτό το μέσο. Από πού θα προέλθουν αυτά τα ευρωπαϊκά χρήματα. Αυτό δεν το είπε ακόμα κανεί, αλλά για μένα δεν μπορεί να είναι μόνο ε, μία ανάληψη από άλλο μέσο ήδη υπάρχουν. Τώρα όσον αφορά τους τοπικούς φορείς, ε, ε, εγώ επιμένω για την επαφή την άμεση. Μου λέτε ναι, μα τα πολιτικά ιδρύματα έχουν ε, μεγάλη εμπειρία κτλ. Και εμείς έχουμε αντιπροσωπείες που βρίσκονται επί τόπου και συμφωνώ απόλυτα, η ΜΚΟ. Τα πολιτικά ιδρύματα που είναι επί τόπου και γνωρίζουν την πραγματικότητα και πρέπει να ωφεληθούμε από αυτήν. Και μάλιστα ο Λάμστορφ είχε προβλέψει και επαφές να ε, μας δώσουν πληροφορίες εντάξει, αλλά για να μετακινηθούν τα κονδύλια και να ανακατανεμηθούν μετά, ε, όχι όμως. Γιατί και πάλι τα πολιτικά ιδρύματα δεν είναι ε, ουδέτερα δεν είναι ουδέτερα ούτε στα κόμματα ούτε στι ε, στις εθνικότητες. Είναι σαφές ότι για τις μικρές χώρες είναι μικρότερα τα ιδρύματα που υπάρχουν, ενώ υπάρχουν και άλλες μεγάλες, ε, μεγάλα ιδρύματα, όπου τα γνωρίζουμε όλοι, είναι τα γερμανικά ιδρύματα. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε πληροφορίες, να συνεργαστούμε μαζί τους, όπως τη ΜΚΟ, η ανοιχτή κοινωνία κτλ. Αλλά Κατά την γνώμη μου και κατά τη γνώμη της ομάδας μου θα πρέπει άμεσα το Ίδρυμα να, ε, να έχει επαφές με τους τοπικούς φορείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η ομάδα των Πρασίνων έχει κάνει αρκετές τροπολογίες στις συστάσεις αυτές. Χαίρομαι που βλέπω να έχουν ενσωματωθεί περισσότερες μία μόνο ε, για την ε, υπηρεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Εκεί θα συνεχίσουμε να αποβάλουμε τροπολογίες. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες. Ε, βέβαια δεν καλύφθηκα εντελώ. Εξακολουθούν να μένουν κάποια ερωτηματικά στο μυαλό μου, ιδίω ό,τι αφορά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Πράγματι, εκεί υπόθηκε ότι πρέπει να γίνουν γρήγορα τα πράγματα για να αναπτυχθεί το έργο του Ιδρύματο. Αλλά νομίζω ξεκάθαρα επίση ε, έλεγαν τα συμπεράσματα ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί συγκεκριμένα τι θα κάνει αυτό το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία και ποια θα είναι η προσθέμενη αξία του. Και αν ε, ισχύουν οι πληροφορίε μου, δεν ξέρω, ο Βιαλίτσκα, ε, κάτι είπε για τα χρήματα. Μήπως ε, έχουν τι τις μεμονωμένες δωρεές περισσότερα χρήματα, τις μεμονωμένες επιδοτήσεις. Αλλά το θέμα είναι ε, αυτό που είπατε για τα καινοτόμα προγράμματα και ιδέες. Θα δώσετε σε ένα μεμονωμένο άτομο τεράστια ποσά και όχι ε, σε κάποιες εταιρείες, απλά και μόνο γιατί είναι καινοτόμο. Το πρόβλημα δηλαδή θα αντιμετωπίσετε κι εσείς τα ίδια προβλήματα με την υπηρεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά τώρα το Open Society, συμφωνώ. Ε, μιλήσατε για την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, έγκυρα τα επιχειρήματά σα, αλλά πρέπει να σα πω ότι αυτή τη βδομάδα σε μια συνάθρηση πολλών κυβερνητικών οργανισμών ακούστηκαν πολλέ προτάσει για το πώ μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση και νομίζω ότι με αυτό το είδημα θα έχουμε βελτίωση. Ελπίζω να καταλήξουμε γρήγορα σε απαντήσεις για όλα αυτά τα θέματα. Επόμενος, ο κύριος Αγκουράκης, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα ευθύ εξ αρχής να ξεκαθαρίσω ότι εγώ τάσουμε ε, με κάθε δυνατή αποφασιστικότητα κατά της ίδρυσης αυτού του ιδρύματος για το οποίο συζητάμε. Ε, και θα έλεγα, μιας και αναφερόμενος και στον τίτλο, να μείνουμε στο ενδεχόμενο, έτσι λέει ο τίτλος, εδώ γίνεται μια συζήτηση λες και έχει αποφασιστεί η δημιουργία του. Και εξηγούμε για ποιο λόγο είμαι τόσο κάθετα αντίθετος. Καταρχήν πρέπει να ξέρετε ότι προέρχομαι από ένα κίνημα το οποίο αγωνίστηκε με όλε τι δυνάμει και σε πολύ δύσκολε συνθήκε για την ανατροπή τη στρατιωτική φασιστική δικτατορία στην Ελλάδα και άρα ξέρω τι σημαίνει να αγωνίζεται κανεί κατά από δύσκολε συνθήκε. Ε, θέλω όμω να πω ότι αυτό το σχήμα το οποίο συζητάτε σήμερα ε, δεν έχει καμία σχέση με την θεμητή πάλι των εργαζομένων και των λαών για δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώματα είναι απλώς ένα φιλοσικής για την προώθηση της υπεριαλιστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άμεση ε, γειτνίασή της και θα κάνει αυτή την πολιτική αν θέλετε ακόμα πιο επιθετική γιατί τώρα βέβαια θα υπάρχει το επιχείρημα ότι τι θέλετε εδώ εμείς χρηματοδοτούμε ε, οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Επίσης κύριε Πρόεδρε δεν είναι τίποτα καινούριο αυτό το Ίδρυμα. Το, ίδιο πράγμα υπάρχει στι ΗΠΑ όπω τα γνωρίζετε. Το έχει ιδρύσει ε, επί εποχή Ρίγκαν και τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ γνωστά. Ένα εκ των οποίων είναι γνωστό επεισόδιο στη Γαλλία μεταξύ του Σοσιαλιστικού Κόμματο και των ΗΠΑ για χρηματοδότηση ακροδεξιού κόμματο. Επίση, νομίζω ότι δεν θέλουν κάποιοι να βγάλουν συμπεράσματα λες και δεν έχουμε ζήσει το, φιάσκο των εγχρώμων επαναστάσεων, των πορτοκαλί επαναστάσεων που έχουν γίνει σε μια σειρά από χώρε, με ολέθριες συνέπειες και μια απαράδεκτη κατάσταση η οποία υπάρχει εκεί. Ε, νομίζω ότι αυτό το Ινστιτούτο θα είναι ένας ε, οργανισμός ανάμειξης ε, στα εσωτερικά των χωρών. Είναι ένα Ινστιτούτο που προωθεί την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως πολύ καλά φαίνεται από την ε, σύσταση των, ε, των ε, governors στους οποίους governors είναι εκπρόσωποι όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης Άρα για ποια ε, ανεξαρτησία από την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μπορεί να ε, μιλάμε. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι δεν θα προσφέρει καμία υπηρεσία, αντίθετα θα αποσταθεροποιήσει την κατάσταση και θα δημιουργήσει ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. κάποια από αυτά τα οποία υπόθηκαν νομίζω ότι δείχνουν ότι υπάρχει επιθυμία για την ίδρυση ενός νέου μέσου. Κάποιοι άλλοι βέβαια λένε ότι δεν θα έχει λόγο ύπαρξη ουσιαστικά αυτό το νέο μέσο. Δηλαδή δεν υπάρχουν ε, στόχοι σχετικά νέοι και υπάρχουν και υποψίες ότι θα μπορούσε να ασκεί παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις κρατών. Αυτό το μέσο, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να ε, λειτουργήσει σε χώρες που δεν υπάρχει δημοκρατία. Ή σε χώρες που είναι πάρα πολύ εύθραυστη η δημοκρατία πρέπει αυτό το μέσο να βοηθήσει την κοινωνία των πολιτών, να στηρίξει αξιόλογες πρωτοβουλίες. Αν συμφωνήσουμε πάνω σε αυτήν την αρχή, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε εύκολα σε ένα συμπέρασμα. Καταλαβαίνω και τις αγωνίες και το άγχος που υπάρχει. Θα πρέπει να ιδωθεί ως ένα συμπληρωματικό μέσο προς άλλα ήδη φυστάμενα μέσα. στην ε, προκαταρκτική αυτή φάση και στην πρόταση Λάμσδορφ, εγώ προσωπικά δεν βλέπω κίνδυνο αλληλοεπικάλυψης με άλλα σχετικά μέσα ή με το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τη Δικαιώματα του ανθρώπου. Πάντως θεωρώ ότι αυτό το νέο ίδρυμα θα πρέπει να προωθεί τη βιώσιμη, την αηφόρο δημοκρατία και να εξακολουθεί να λειτουργεί εκεί που η δημοκρατία είναι πάρα πολύ εύθραυστη. Να χρησιμοποιείται με έναν τρόπο που να μην παρεμβαίνει, απλά να μπορούν να επωφεληθούν από αυτό όσο δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι και ταυτόχρονα θα πρέπει να μπορεί να διοχετεύει άμεσα τα κονδύλια στους δικαιούχους. Ο κύριος Βιαλίτσκα πολύ ξεκάθαρα μας είπε πού βρίσκονται οι κίνδυνοι. Έχουμε την ε, περίπτωση Άλες Μπιαλέσκη που ήρθε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και μας ε, μίλησε. Και είναι ένα παράδειγμα του κινδύνου ε, που μπορεί να ελοχεύει με την υπερβολικά μεγάλη διαφάνεια. Δηλαδή ε, μπορεί να έχει κάποιος αντίπεινο να υποστεί αν έχει λάβει κάποια κονδύλα, κάποια βοήθεια. Πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί λοιπόν στον τρόπο από τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο μέσο. Θα πρέπει με έναν γρήγορο, αλλά θα πρέπει να γίνεται και διακριτική χρήση της χρηματοδότησης. Ευχαριστώ. Κόβαλ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή μας δείχνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε για να ιδρυθεί αυτό το ίδρυμα, γιατί πολλοί περιμένουν Δεν φαίνεται όμω στον προπολογισμό του 2012 αυτό το, νέο μέσο. Μιλάμε για 96 δις ευρώ για κάθε είδους προγράμματα, τίποτε όμως για το Ευρωπαϊκό Δήμα για τη Δημοκρατία. Γιατί, ερωτώ. Σε ό,τι αφορά τώρα τους νέους. Η κατάσταση επιτόπου έχει αλλάξει. Η κατάσταση προ και μετά εκδημοκρατισμό είναι διαφορετική. Δηλαδή βλέπουμε νέους ανθρώπους να δυσκολεύονται στη ζωή τους. Να δυσκολεύονται και με το κράτος, στις ε, δοσοληψίες με το κράτος. Αλλά είναι μια ομάδα που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, να τη δούμε ω συνομιλητή. Τι είπε και ο κύριος Πέτερινγκ, το Ίδρυμα Κοντράντ Αντενάουερ και ο κύριος Πέτερινγκ είναι πολύ θαραλέοι και τολμηροί. Χρειάζονται οι αρέτες αυτές, γιατί ο εκδημοκρατισμός δεν γίνεται αν δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να στηρίζουμε τη δημιουργία νέων πολιτικών κομμάτων, αλλά χωρίς να παρεμβαίνουμε πολιτικά, γιατί αρκετά δύσκολη είναι η πολιτική στη διαδικασία μετασχηματισμού. Πρόεδρος, επειδή ήταν πάρα πολύ ζωντανή και έντονη η συζήτηση, αλλά πρέπει να διακόψουμε και για τις, τους διερμηνείς, θα ήθελα να δώσω στην υπηρεσία δράση ε, το λόγο εν συντομή για να δώσει κάποιες απαντήσεις για θέματα τα οποία προέκυψαν και μετά να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ποπόφς και δυστυχώς δεν έρχεται γιατί εκλήθη επιγόντως σε μια συνάντηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και δεν μπόρεσε να έρθει εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω ε, τον Αλεξάνδρ Λάμστρομ για την εξαιρετική του πρόταση και να ευχαριστήσω και τους κοιόδης εισηγητές εκ μέρους της εξωτερικής δράσης για τη θετική ανάλυση και τη θετική τους ανταπόκριση στην πρόταση που έχουμε επιτάπητος. Χαίρομαι γιατί βλέπω ότι φαίνεται να κινούμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και αυτό πρέπει να το εκφράσουμε με ικανοποίηση. Εγώ νιώθω μεγάλη προσμονή για αυτή την πρωτοβουλία και το ίδιο ε, διαστάνομαι ακούγοντα του συναδέλφου με το πάνελ. Όλα αυτά είναι ένα σαφέ ε, δείγμα του πόσο απαραίτητο είναι αυτό το νέο μέσο, γιατί πρέπει να καλύψουμε κάποια κενά. Και το είδαμε και πολύ έντονα νωρίτερα φέτο, όταν προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε με τον κατάλληλο τρόπο τι αλλαγέ στη Βόρεια Αφρική. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, ναι, θα συνεχίσουν οι εργασίε, ναι, χρειάζονται περισσότερε λεπτομέρειε και όπω ανέφερα, η ομάδα εργασία ε, θα συγκροτηθεί, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει αν δεν συμμετέχει σε αυτές τις εργασίες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποια πιο συγκεκριμένα θέματα στη διάρκεια της διαδικασίας. Επίσης, πολύ σημαντικό ήταν ο ρόλος του Κοινοβουλίου και σε αυτό το νέο ε, σχηματισμό, σε αυτήν την ομάδα εργασίας, αλλά και ε, ως φορέας κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, το Ίδρυμα ποτέ δεν ε, θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να πάρει πόρους οι οποίοι ε, πηγαίνουν σε αυτό το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, γιατί είναι ένα μέσο πολύ σημαντικό για όλους μας. Δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε τον τρόπο λειτουργίας του. Υπάρχει ένα κενό όμως που δεν μπορεί να το καλύψει αυτό το ευρωπαϊκό μέσο. Ούτε βλέπουμε τρόπο να αυτομεταρρυθμιστεί και δεν μπορεί να ασχοληθεί με όλα όσα ε, θα πρέπει να αποτελούν αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού για τη Δημοκρατία. Το θέμα είναι ε, να μην υπάρχει σύγχυση μεταξύ δικαιούχων και αποδεκτών. Ουσιαστικά δίνουμε κάποιους ε, πόρους, κάποιο αρχικό κεφάλαιο, αν θέλετε, σε κάποιους που θέλουν να οργανωθούν και να δημιουργήσουν συνθήκες για περισσότερο πλουραλισμό, μεγαλύτερη δημοκρατία, Άπαξ και οι πρωτοβουλίε αυτέ λάβουν σάρκα και οστά, δεν ξέρω αν είναι πολίτε, δημοσιογράφοι, οτιδήποτε. Έπειτα αυτοί θα μπορούν να είναι επιλέξιμοι για την χρηματοδότησή του είτε από το Ευρωπαϊκό Μέσο, είτε Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ή για οποιοδήποτε, από οποιοδήποτε άλλο μέσο. Άρα δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Εμεί στηρίζουμε μόνο τη σύσταση. Άρα υπάρχει προστέμινη και συμπληρωματικότητα. Τώρα, τέλος, διαβουλεύσεις και συνεργασία με άλλους φορείς, μη κυβερνητικέ οργανώσεις και ε, πολιτικά ιδρύματα. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ απαραίτητο και σημαντικό όσοι έχουν εμπειρία ε, σε ό,τι αφορά την παροχή υποστήριξη ε, σε χώρες που βρίσκονται σε μετάβαση μπορούν να μας βοηθήσουν και μπορούμε να διδαχθούμε πολλά από αυτούς. Ο πρόεδρο, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η ανακεφαλαίωση αυτή. Θα κλείσω τη συνάντηση εκφράζοντα ευχαριστίε μου προ τη Γραμματεία και το προσωπικό που οργάνωσαν αυτή την ακρόαση και που εξακολουθούν να επεξεργάζονται τι προτάσει για, για αυτή την πρόταση. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με του συναδέλφου και να πω δύο πράγματα εν κατακλείδη. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για τη σύσταση 15 Δεκεμβρίου την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Και επίση οποιαδήποτε γραπτή τροπολογία θα πρέπει να έχει πριν από αυτή την ημερομηνία. Επόμενη συνεδρίαση, Δευτέρα 6.30 το απόγευμα στο Στρασβούργο είναι η επόμενη συνεδρία, παρουσία της Αντιπρόεδρου της Κομισιόν και είπα εκπροσώπου. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και όλες. Γεια σας.